Πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ. Είναι έξι τα επιμέρους ψηφίσματα. Πρώτος ο μιλητής, ο Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, για έναν Ισπανό το να πρέπει να κακολογήσει μία χώρα όπως η Βενεζουέλα είναι οδυνηρό. Γιατί έχουμε ε, μακραίων ιστορικούς και πολιτισμικούς ε, ε, θεσμούς και πολύ θερμά αισθήματα που δεν θα αλλάξουν ποτέ. Αλλά έχουν πάει πολύ μακριά τα πράγματα. Οι δύο σημαντικότερες ομάδες ε, αντιπολίτευσης ε, κατέληξαν εδώ σε μια πολύ ρητική κατηγορηματική και στεναρή ε, πρόταση ψηφίσματος που καταδικάζει δρυμύτατα την πολιτική του Πρόεδρου Μαδούρο. Γιατί ασκούνται διώξει κατά της αντιπολίτευσης και μάλιστα η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε ε, την ε, Βενεζουέλα ως χώρα χωρίς ελευθερία έκφρασης, χωρίς ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ε, χώρα που εφαρμόζει βασανιστήρια. Όλα αυτά δεν είναι απλά λόγια. Μέχρι πότε θα χρησιμοποιεί και θα εκμεταλλεύεται την υπομονή μας ο κύριος Μαντούρο και θα χρησιμοποιεί την ομοποίηση του και τη δημοκρατική του εκλογή για να ε, προσβάλλει έναν ε, πρώην πρόεδρο, τον κύριο Αθηνάρ, καταδικάζοντας τον ως πραξικόπηματία ενώ ο ίδιος είναι επίγονος πραξικοπηματία. Ευχόμαστε για τη Βενεζουέλα ευημερία, δημοκρατική πορεία, ειρήνη και ελπίζουμε να βρει ένα δρόμο ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τη χώρα αυτή για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2013 η κατάσταση επιδεινώθηκε τραγικά στη Βενεζουέλα. Για την αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ε, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται συλλήψεις. Ε, ε, η σύλληψη του ηγέτη της αντιπολίτευση Λόπες ήταν βέβαια το αποκορύφωμα. Ο ύπατος αρμοστής ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση και διαπίστωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών. Η χώρα είναι διχασμένη ε, το ρήγμα ε, διαχωρίζει ακόμα και οικογένειες. Η παρούσα κυβέρνηση της Βενεζουέλας πρέπει λοιπόν να κλείσει αυτό το δυσάρεστο κεφάλαιο και να ξεκινήσει τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση. Κυρίως οι Αθώοι θα πρέπει να αφαιθούν πάρα αυτά ελεύθεροι, να υπάρχει διασφάλιση του δικαιώματος ε, του συνέρχεστε και να επανέλθει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμασμάκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προσυπογράψω τα όσα αναφέρθηκαν από τους προραλήσαντες συναδέλφους Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση και ο πρόεδρος Μαδούρο ε, και η κυβέρνησή του προσπαθούν ε, βία ε, να σταματήσουν τις διαδηλώσεις. Έχουν μπει στις φυλακές 1.400 άτομα. Έχει δυσκολέψει η πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο πρόεδρος ε, Μαδούρο συνέχισε την πολιτική του πρόεδρου Τσάβες ε, και ε, προχωράει με, μια, με ένα κληροδότημα το οποίο έχει οδηγήσει σε πληθωρισμό 60% σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ενδεχομένως ίσως θα πρέπει να ασκήσουμε κυρώσεις και πιέσεις κατά της κυβέρνησης Μαδούρο και ενδεχομένως ε, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα να μην έχουν πλέον πρόσβαση στο ε, έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάσουμε απερίφραστα τις παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Βενεζουέλα. Ευχαριστώ κύριο Κοράο όσον αφορά το θέμα της ε, ε, Βενεζουέλας, όπως συχνά γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, στη διάρκεια ε, της συζήτησης είχα την αίσθηση ότι το πρόβλημα δεν είναι πραγματικό, αλλά ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι με φανατισμό το αντιμετωπίζουν δεν καταφέρνουμε να δούμε τα πράγματα με πραγματικά αντικειμενικό τρόπο. Από τη μία πλευρά έχουμε τους υποστηρικτές του Προέδρου Μαδούρου, Μαδούρο, ε, τους φιλοκυβερνητικούς δηλαδή, και από την άλλη πλευρά αυτούς που στηρίζουν την αντιπολίτευση, που όμως ε, ενδεχομένως ε, δεν είναι αυθόρμητη αντιπολίτευση, αλλά υποκινείται από κάποια άλλη εξωτερική δύναμη. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα αντικειμενικά. Να βρούμε οργανισμούς οι οποίοι ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν ε, τον πληθυσμό της Βενεζουέλας ε, και να κυδεμονεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το ψήφισμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο και μπορώ σήμερα να πω υπερήφανο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και σε μια ιστορική στιγμή κατάφερε να ανταποκριθεί με κατηγορηματικό και στεναρό τρόπο στην έκκληση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Παρ' όλα αυτά και παρά τη στεναρότητα του, ψηφίσματο ψηφίσματός μας, δεν θα πρέπει να υποπέσουμε στο σφάλμα και να θεωρήσουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θα πρέπει από το ψήφισμα αυτό και μετά να συνεχίσουμε τι προσπάθειές μα, ώστε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διορθώσει, αν γίνεται, και να σταματήσει την κατάφορη παραβίαση και συστηματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιδών ελευθεριών των πολιτικών αντιφρονούντων. Αν δεν γίνει αυτή η διόρθωση, σας διαβεβαιώ εκ μέρους των φιλελευθέρων ότι θα διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει τη συμπεριφορά τη. Σα ευχαριστώ, κύριο Κόουζο. Μερικοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τους βολεύει και όπως τους συμφέρει. Το ψήφισμα αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής κατήχησης και χειραγώγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, γιατί ε, ο λαός της Βενεζουέλας ε, διάλεξε ελεύθερα το δρόμο του και παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε πραξικοπήματα, πετρελαϊκό σαμποτάζ, χειραγώγηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εδώ βλέπουμε, βλέπετε εδώ ειρηνικού διαδηλωτέ, ε, βλέπουμε όπλα στις φωτογραφίες, βλέπουμε ρήψει ε, ε, όπλων και όλμων. Επίσης, 11 ε, αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στη Βενεζουέλα και μάλιστα ενώ στην Ισπανία έχουμε νόμους που απαγορεύουν τις, στις διαδηλώσεις, ε, απαγορεύουν τις διαδηλώσεις. Παρ' αυτά δεν επιτρέπουμε κάτι τέτοιο στη Βενεζουέλα και ουσιαστικά δεν επιτρέπουμε τον βενεζουελικό λαό να ε, διαλέξει ελεύθερα την πορεία του. Ευχαριστώ κύριο Στετίνα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το καθεστώς ε, της ε, Βενεζουέλας προσπαθεί να φημώσει την ε, αντιπολίτευση και πολλοί χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταλήξει στις φυλακές μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και πολιτικοί όπως ο Λεοπόλντο Λόπες και ο Ντανιέλ Θεβάγιος. Ε, γνωρίζουμε την ε, ιστορία της ε, χώρας αυτής και εμείς την καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο γιατί προερχόμαστε από σοβιετικά καθεστώτα. Γνωρίζουμε τι σημαίνει δίωξη, πολιτική δίωξη, εγκλισμός σε φυλακές και επομένως θα πρέπει να ξανακάνουμε αυτό που έγινε προς εμάς τόσα χρόνια πριν, δηλαδή στήριξη από την πλευρά των δημοκρατικών χωρών. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ε, ζητώ άμεση απελευθέρωση του Λεοπόλντο Λόπες και άλλων πολιτικών κρατουμένων. Ευχαριστώ. Ασίς. Ο κύριος ασίς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια δημοκρατία κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να αποσυνδέεται από το κράτος δικαίου και κράτος δικαίου προϋποθέτει θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Καταρχήν διάκριση των εξουσιών, σεβασμός της ατομικής ελευθερίας και της ελευθερίας έκφρασης. Και ο σεβασμός ε, του κράτους δικαίου εξασφαλίζεται πάνω απ' όλα από την κυβέρνηση μιας χώρας. Και γι' αυτό οι σοσιαλιστές ε, ε, συνέβαλαν τα μάλα στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Είμαστε κατά της πιθανότητας επιβολής κυρώσεως στη χώρα αυτή. Είναι υπερβολικό και δεν έχει καμία σχέση με η σημερινή κατάσταση στη Βενεζουέλα με αυτά που συνέβησαν στη Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή. Και φυσικά θα πρέπει να έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να διαδηλώνει ειρηνικά, κάτι που δεν συνέβη πάντα. Εμεί είμαστε υπέρ τη πρόταση, συμμετείχαμε στην εκπόνηση του ψηφίσματο αυτού, γιατί πάνω απ' όλα προέχει ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν την Βενεζουέλα, γιατί όντως εμφανίζονται κάποιε καταστάσεις που καταπατούν αυτή την αρχή αλλά πρέπει να κάνουμε μια γενική αναφορά της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα είναι κατά τη γνώμη μας μια δημοκρατική κοινωνία, γίνονται εκλογές. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατική κοινωνία της Βενεζουέλας έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει πλήρως το λόγο του και να βοηθήσει. Ευχαριστώ. Μία μπλε κάρτα από την κυρία Βεσέρα έχει υποβληθεί κυρία Σεις. Θέλετε να την ακούσετε, κυρία Βεσέρα. Θα ήθελα να προσθέσω απλώς κάτι και να πω ότι αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Βενεζουέλα και σχετική συζήτηση είναι πολύ σημαντική και αποφασιστική σημασία. Ουσιαστικά συσπηρωνόμαστε και συνενώνουμε τις δυνάμεις μας, αλλά δεν τονίζουμε δεόντως κάτι που είναι πολύ σημαντικό, που είναι η πολιτική δίωξη που λαμβάνει η χώρα. Ποια είναι η ερώτηση σας κυρία Μπεσέρα, γιατί η μπλε κάρτα προϋποθέτει ερώτηση. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, θα επιμείνουμε ώστε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Βέλγιο που αναγνώρισε ως τούντες σε πολιτικό άσυλο κατοίκους της Βενεζουέλας να συνεχίσει και να μην λαμβάνει υπόψη αυτή την πολιτική δίωξη. Ο κύριος Ασίσου. Η ψηφοφορία που θα γίνει εντό ολίγου και το υπερψήφι, υπερψήφιση ακριβώ του ψηφίσματο ουσιαστικά αναγνωρίζει κάποιε καταστάσει ε, που χρήζουν ε, στηλίτευση, όπω η κατάσταση που λαμβάνει η χώρα στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή και που παραβιάζει και ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κάτι όμω που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια στη Βενεζουέλα γίνονταν δημοκρατικέ εκλογέ. Βέβαια αυτό δεν αρκεί για να εδραιωθεί πλήρω μια δημοκρατία. Μια δημοκρατία δεν περιορίζεται στι εκλογικέ αναμετρήσει. Η δημοκρατία προϋποθέτει σεβασμό των αρχών του κράτου δικαίου. Και όταν διαπιστώνουμε παραβίαση θα πρέπει να το δηλώνουμε. Ευχαριστώ. Κύριο Κάρσκι. Κύριε Πρόεδρε. Ε, τον Φεβρουάριο συνελήθησαν φοιτητέ υπό το, το πρόσχημα της υποκίνησης ε, ε, δια, διάπραξη εγκλήματος, ενώ ήταν ειρηνικοί διαδηλωτές. Επίσης, ο κύριος Λόπες ε, κατηγορήθηκε από τις αρχές Βενεζουέλας για υποκίνηση διαδηλώσεων η δικαστική εξουσία δεν είναι δίκαιη και ουσιαστικά προσάγει στη δικαιοσύνη ε, ειρηνικούς διαδηλωτές. Οι συλλήψεις, κρατήσεις ε, και του Λεοπολδολόπης και άλλων είναι παράνομη πράξη, αδικαιολόγητη και παράτυπη. Δεν ε, ε, είναι σωστή αυτή η εξευθυλιστική, ταπεινωτική και αντιδημοκρατική αντιμετώπιση των δημοκρατικών δυνάμεων. Παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν η διεθνή κοινότητα να αναλάβει κάποια δράση κατά του καθεστώτος του Νικόλα Μαντούρο για να εξασφαλιστεί η τήρηση ε, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και θεμελιδιών ελευθεριών στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαλάντσοβα γινόμαστε μάρτυρες μια σοβαρής επιδείνωσης των δικαιωμάτων των, του λαού της Βενεζουέλας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση και να οξυνθεί. Γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο να εξετάσει ακόμη και την επιβολή συγκεκριμένων κυρώσεων προς συγκεκριμένους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο. Ε, βλέπω με αποτροπιασμό το πώς η κυβέρνηση και το καθεστώς αντιμετωπίζει τους πολίτες. Άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά, που ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα κατά της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής, εκτίθενται σε καταστολή, σε βιοπραγία και συστηματική άσκηση, βία, άσκηση βίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων που συνελήθησαν με αυθαίρετο τρόπο, παράνομα και χωρίς να έχουν δικαίωμα δίκης μεταχείρισης, μεταξύ άλλων του Λεοπόλτο Λόπες και της Μαρίας Ματσάδο. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αρχηγοί της αντιπολίτευσης να υφίστανται πολιτικές διώξεις και να τιμωρούνται ενώ η δικαστική εξουσία δεν είναι λειτουργική στη Βενεζουέλα, ούτε είναι ανεξάρτητη, ώστε να μπορεί να διερευνά και να κρίνει με δίκαιο τρόπο τέτοιου είδους καταστάσεις. Ευχαριστώ κύριο Χρυσόγωνος. <clears throat> Αφετηρία των αιματηρών συγκρούσεων φέτος στη Βενεζουέλα ήταν η προσπάθεια της άκροδεξιάς να ανατρέψει με τη βία τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση Μαδούρο. Αντί λοιπόν οι κυρίαρχες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικές δυνάμεις να εγκαλούν την κυβέρνηση της βενεζουέλας χρησιμοποιώντας μάλιστα κατά επιλεκτικό τρόπο στοιχεία από την έκθεση του επιτετραμένου των ηνωμένων εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλ χουσέιν καλύτερα θα έκαναν να ασχοληθούν με την αντίστοιχη έκθεση του επιτετραμένου, των ηνωμένων εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σέφας λούμινα η οποία διαπιστώνει συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελλάδα του μνημονίου εξαιτία των πολιτικών εξοντωτικής λιτότητας που επιβάλλουν η τρόικα και το εκοφίν. και αντί για μαθήματα δημοκρατίας στη βενεζουέλα καλύτερα θα έκαναν να δείξουν μεγαλύτερο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες στα κράτη μέλη της ένωσης και να σταματήσουν τις προσπάθειες εκβιασμού συνειδήσεων ελλήνων βουλευτών και ψηφοφόρων με τις απειλές περί χρεοκοπίας εξόδου από την ευρωζώνη και άλλα παρόμοια που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες. <clears throat> Κύριε Χρυσόγονε, έχετε μία ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Μπούχνερ. Θέλετε να την δέχεστε να την λάβετε. Κύριε Μπούχνερ, παρακαλώ. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι στη Βενεζουέλα η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τη βία, την παρανομία όμως από την άλλη ισχύει επίσης ε, ότι ε, δεν ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα βασανιστήρια και θα θέλω να απαντήσετε από αυτού παρακαλώ. Terror und Κοιτάξτε, η τρομοκρατία ε, και τα βασανιστήρια προφανώς και δεν αιτιολογούνται από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται. Όμως στην περίπτωση αυτή έχουμε διαδικασίες νομότυπες ε, κατά ανθρώπων που πράγματι υπέστησαν ή διέπραξαν εγκληματικές πράξεις στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Ουρτάσουν. Ε, εγώ νομίζω ότι εδώ χρησιμοποιούμε άσχημα το άρθρο 135 γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε ε, για γενικά κατά μιας ε, ενώ μιλάμε για συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, νομίζω ότι ε, δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Από τη μία δηλαδή να χειροκροτούν καθεστώτα πολύ δικτατορικά και από την άλλη να κάνουν αυτή τη συζήτηση για την Βενεζουέλα. Δεν είναι δυνατόν να γενικεύουμε είναι σε καταστάσει. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την υποκριτική στάση. Εμεί δεν θέλουμε ούτε να, συζητήσουμε, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση, ούτε να υποβάλουμε ε, τροπολογίε και οπωσδήποτε θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ουρτάσουν, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρσκι. Τη δέχεστε? Παρακαλώ κύριε Κάρσκι. padło τέτοιο είδους ε, ε, υποτιμητικά σχόλια είναι απαράδεκτα. Ε, δέχεστε δηλαδή τις εξευτελιστικές συμπεριφορές κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Λεοπόλτο Λόπες και άλλων συλληθέντων ακτιβιστών της αντιπολίτευσης. Τους έδειξαν περιτώματα. Είναι ταπεινωτική εξευτελιστική αυτή η συμπεριφορά. Είναι απαράδεκτο. Επίσης Ταυτόχρονα ακούμε τους ε, ύμνους ε, ε, που με εκοφεντικό τρόπο ηχούν στις φυλακές και βασανίζουν τους πολιτικούς κρατουμένους με συνθήματα όπως ο Τσάβες ζει, ο αγώνας συνεχίζεται. Συμφωνείτε με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ απλώς λέω ότι θέλω ίδια μέτρα και σταθμά για όλες τις χώρες. Ε, ε δεν είναι δυνατόν εδώ να κάνουμε μια γενική δίκη κατά μιας ε, κυβέρνησης. Ε, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβιάσεων και να τις συζητήσουν. Εδώ έχουμε 8 ψηφίσματα για την Βενεζουέλα, οι οποίες περιεχόμενο έχουν απλώς κατά της κυβέρνησης να γίνονται συζητήσεις. Άλλη μια μπλε κάρτα από τον κύριο Βάρτη από τον κύριο Νάρτ. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Νάρτ, παρακαλώ. Σύντροφε Ουρτασούν, θεωρείτε λογικό ο εισηγητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και ο εισηγητής ε, τη Επιτροπής κατά των βασανιστήριων των Ηνωμένων Εθνών ε, και άλλοι αντίστοιχοι οργανισμοί ε, να συζητούν τέτοια πράγματα και η, δυνατότητα, η μη δυνατότητα προσφυγής στο Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων ε, του Ανθρώπου από πλευράς ε, των πολιτών της ε, Βενεζουέλας είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να καταδικαστούν. Εγώ το λέω για όλες τις περιπτώσεις. Εγώ το λέω για όλες τις περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές είναι συγκεκριμένε περιπτώσεις και πρέπει να τις καταδικάσουμε. Δεν καταδικάζουμε αυτά που δεν είναι καταδικαστέα, καταδικάζουμε αυτά που είναι καταδικαστέα. Javier, no es eso. Yo voy a... Yo φυσικά θα ε, στυλιτεύω την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και λαμβάνω χώρα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, Χαβιέρ. Εδώ πρόκειται για κάτι γενικό. Έγιναν άπειρα ψηφίσματα για τη Βενεζουέλα, γιατί έχουμε κάποιους ευρωβουλευτές ε, που θέλουν να κάνουν ε, κήρυγμα και έχουν πραγματικά μένονται λισαλέα κατά της Βενεζουέλας. Έχουμε πολλές μπλε αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και, άλλο δύο συζητήσεις, και άλλες δύο συζητήσεις για άλλα δύο κατεπήγοντα. Γι' αυτό πολύ λυπούμε, αλλά δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ετούντες μπλε κάρτα. Και θα είμαι πολύ πιο αυστηρός από εδώ και πέρα στην τήρηση του χρόνου. Γιατί θα καθυστερήσουμε αν δεν τηρήσουμε όλη του χρόνο αγόρευση. Ο κύριος Μπασίρ. Uh, Mr. President, Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να καλέσω την κυβέρνηση Ομπάμα να ξεκινήσει το διάλογο με τη Βενεζουέλα ακριβώς όπως έκανε και με την Κούβα. Ε, ας μην χρησιμοποιούμε πλέον ε, προσχήματα του καθεστώτος της Βενεζουέλας ε, χρησιμοποιούνται για να περιοριστούν η ελευθεροτυπία, ε, για να παρεμποδιστεί η πραγματική δημοκρατία και για να εφαρμόζονται κατασταλτικά μέτρα. Όταν η Βενεζουέλα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί πλέον να στηρίξει την οικονομία της γιατί ανά τον κόσμο ε, πέφτει η τιμή του πετρελαίου πλέον το 60%, μάλλον ο πληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα ανέβει στο 60% και δεν θα μπορεί πλέον η Βενεζουέλα να προσφέρει στους πολίτες της όλα αυτά που τους έχει υποσχεθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ακριβώς όπως έγινε και με την Κούβα, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να καταπιέζουν τις φιλοδοξίες ε, ενός άλλου ε, κυριαρχού κράτου. Σα ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλου του παριστάμενου ευρωβουλευτέ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη καινούργια χρονιά. Ευχαριστούμε κύριε Μπασίρ. Ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ βαθύτατα για τη συνεχή επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα έχει ευθύνη και υποχρέωση να πληρεί τις διατάξεις του κράτους δικαίου, γιατί μόλις έγινε και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ε, του ΟΗΕ. Αντίθετα, έχουμε αυξανόμενη ιδεολογική και πολιτική αδιαλαξία ε, και μυσαλλοδοξία Είχαμε την σύλληψη του αρχηγού της αντιπολίτευσης Λόπες και επίσης ε, σκανδαλώδη αποπομπή γερουσιαστών και οι ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από παραστρατητικές φιλοκυβερνητικές δυνάμεις ένοπλες. Εκφράζουμε την συμπαράσταση και την ελληνική μας προς το λαό και τους ακτιβιστές που προσπαθούν να επαναφέρουν τη Βενεζουέλα στο δρόμο της δημοκρατίας και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυρία Μαγκερίνη να ζητήσουν την άμεση άμεση αποφυλάκηση των διαδηλωτών και των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πέραν ε, των άστοχων διατυπώσεων και ίσως τη μεροληψία κάποιων παραγράφων του ψηφίσματος είναι σίγουρο ότι όλοι οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες της Βενεζουέλας θα πρέπει να συμβάλλουν και να συμμετέχουν σε έναν διάλογο που πρώτα απ' όλα θα έχει την άμεση κατάπαυση της βίας και την έναρξη ενό διαλόγου που θα επιτρέψει την ειρήνη και θα επαναφέρει την ελευθερία του συνέρχεστε και του συναθρίζεσαι χωρίς άσκηση βίας θα πρέπει να αφήσει τις αυθαίρετες ε, ενέργειες, όπως τις αυθαίρετη κράτηση του Λεοπόρντο Λόπελς, που εδώ και μήνες ε, ε, είναι φυλακισμένος από, είναι φυλακισμένος από παρόλο που η κράτησή του έχει κηρυχθεί ε, αυθαίρετη από πολλές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστήριων, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί η διάκριση των εξουσιών στη Βενεζουέλα. Είναι αδύνατο να κρατείται κάποιος σε μια στρατιωτική φυλακή για ένα θέμα που σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει σε στρατιωτική δικαιοδοσία. Επίσης, ε, αυτή τη στιγμή η βασική σύγκρουση της Βενεζουέλας δεν είναι ε, μεταξύ ε, σοσιαλιστών και καπιταλιστών. Είναι μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι η βία είναι πολιτικό εργαλείο και εκείνων που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για να εμποδίσουν μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπέλντερ. Μια φράση έχω να πω. Η δημοκρατική αντιπολίτευση στην ε, Βενεζουέλα δεν έχει κανένα δικαίωμα, δεν μπορεί να μιλήσει. Μας λένε στην Βενεζουέλα ότι η χώρα έχει ε, εκδημοκρατήσει την παρανομία ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε την δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας που επιθυμεί την, ε, το κράτος δικαίου και την αποκατάστασή του δεν είναι δυνατόν ε, να ε, βλέπουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες κατά τις ε, και κινήσεις κατά τις αντιπολίτευσης οι οποίες συνοδεύονται και από κινήσεις αντισημιτισμού. <clears throat> Αυτό είναι απαράδεκτο και ήθελα να το πω γιατί κανείς δεν το έχει αναφέρει. Η κυρία Μπέβερ σήμερα Στη Βενεζουέλα ε, πολλοί από τους ε, ηγέτε τη αντιπολίτευση βρίσκονται στη φυλακή. Ο κύριο Λόπε είναι ο πιο γνωστός, αλλά περίπου 100 εκτιβιστές και αυτοί βρίσκονται στη φυλακή. Πάνω από 2.000 ε, εναντίον του κρεμούν υποθέσει, βρίσκονται υπό ανάκριση και Όλοι αυτοί θέλησαν να διαμαρτυρηθούν κατά τη κυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα στο χείλο ε, τη καταστροφή. Ο κύριο Μαντούρο οφείλει να κατανοήσει ότι στη δημοκρατία ε, μπορούμε να διαπραγματευόμεθα με του ε, αντιπάλου μα. Δεν του βάζουμε στη φυλακή, δεν τερματίζουμε με αυτόν τον τρόπο ούτε τη ζωή του ούτε την σταδιοδρομία του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να απελευθερωθούν πάρα αυτά οι πολιτικοί κρατούμενοι, να καταργηθούν τα βασανιστήρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την απελευθέρωσή του. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να πιστεύουμε όλοι ότι εδώ υπάρχει συνωμοσία κατά τη Βενεζουέλας. Το αντίθετο ισχύει. Εμεί θέλουμε η Βενεζουέλα να ακολουθήσει το δημοκρατικό δρόμο οι άνθρωποι να ζουν με ασφάλεια και ευημερία. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Ζουμπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βιαιότητες, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, ε, εμπρισμός νηπιαγωγείων, νοσοκομείων και μάλιστα ένα μωρό έχασε τη ζωή του στον εμπρισμό ε, ενός νηπιαγωγείου και γιατί η διαταγή ήταν να ε, κάψτε παντού. Αυτά είναι πολύ σοβαρά εγκλήματα σε όλες τις χώρες ε, και αυτοί που οργάνωσαν αυτά τα εγκλήματα ή τα υποκίνησαν στις δικές μας χώρες θα, θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Στην Βενεζουέλα όμως τα θύματα δεν είναι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτοί που προκάλεσαν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Αυτό δεν το αναφέρεται όμως. Αυτή τη στιγμή έχουμε 34 άτομα στη Βενεζουέλα που έχουν διαπράξει σοβαρότητα εγκλήματα που και 14 ε, άτομα της αστυνομία που κατηγορούνται για, για υπερβολική χρησιβία. Θα πρέπει να μην εθετούμε διπλά μέτρα και σταθμά και σίγουρα όχι νεοαπικιοκρατική συμπεριφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ακριβώς το ψήφισμα αυτό συνιστά την έκφαση χειραγώγησης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από εξτρεμιστικές δυνάμεις της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όμως όλους τους ε, ομιλητές γιατί επαναλαμβάνω πρέπει να διεκπαιρεώσουμε εγκαίρως και τις υπόλοιπες συζητήσει. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο μόνο σε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα και εφόσον δεν έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Ο κύριος Τουργκάης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι κατεπίγουσα και μάλιστα διεθνώ. Ε, η κυβέρνηση Μαντούρα που συνεχίζει το, το καθεστώ του Τσάβε ε, είναι δικτατορική κυβέρνηση. Θέλει να φημώσει την αντιπολίτευση, ε, να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενισχύσει του τρομοκράτε και να καταστήλει και να καταπιέσει, να φτωχύνει το, το λαό τη Βενεζουέλα. Είναι μια δημοκρατία φρίκη όπου συλλαμβάνονται και φυλακίζονται όσοι είναι κατά του Μαδούρο και όσοι δεν ε, ε, εστερνίζονται το δόγμα του Τσάβες. Καταπιέζεται και διώκεται ο λαός της Βενεζουέλας από τους ε, εξτρεμιστές του Τσάβες. τέλειωσε ο χρόνος για τα λόγια, πρέπει να περάσουμε στα έργα. Θα πρέπει να σταματήσει την αντιδημοκρατική κλιμάκωση που έχει ξεκινήσει η Βενεζουέλα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η Βενεζουέλα θα ξυπνήσει από αυτόν τον εφιάλτη του Τσάβες και θα γίνει μια πραγματικά δημοκρατική χώρα με ελευθερίες και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει μάχη για να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Και όσοι είναι υπέρ ε, του Τσάβες, της, του, ε, παρόμοιο του Τσάβες της Βενεζουέλα, όπως το Ποδέμος του κυρίου Ιγλέσιας, ε, με δηλία ε, έλαμψε δια της απουσίας του και δεν τόλμησε να έρθει και να πει τίποτα κατά της κυβέρνησης Μαδούρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, έχει δράσει σε διεθνές επίπεδο υπέρ της δημοκρατίας και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και επομένως εμείς δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπέρ ε, των διαδικασιών, των δικαίων διαδικασιών. Ε, επομένως πραγματικά είναι μέσα στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για την κατάσταση στη Βενεζουέλα όπου καταπατούνται διαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στηρίζουμε το ψήφισμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεταφέρει αυτό το μήνυμα για ανάγκη κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων και σεβασμού των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν αυτές οι καταχρηστικές ε, καταστάσεις. Ε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα πρέπει να κάνει πραγματική ε, πρόοδο, να επιτρέψει το συνεταιρίζεστε, να επιτρέψει την ελευθερία του λόγου και τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί από όλους τους φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει, είπα, η εκπρόσωπος να παίξει σημαντικότερο ρόλο. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα, ήλπιζα να μιλήσω για να επισημάνω την περίπτωση της κυρίας Ματσάντο, αλλά τώρα θα μιλήσω με βάση τα σχόλια που έγιναν, ε, με βάση αυτά που είπε χθες ο πρέσβης ε, στην αντιπροσωπεία για τη Μερκεσούρ και είπε ότι ο κύριος Λόπες ε, είναι υπέτειος, φταίει, έχει διαπράξει εγκλήματα και είπε ότι θα υπάρξει δίκαιη δίκη. Αυτό όμως είναι παράλογο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρξει δίκαιη δίκη στη Βενεζουέλα, αυτό νομίζω είναι απόλυτα σαφές. Το καθεστώς είναι εκτεθειμένο και θα ήταν κομικό να μιλάμε για δίκαιη δίκη γιατί παράλληλα βλέπουμε ότι οι απλοί πολίτες ζουν στη φτώχεια η ακρά ειδιστερά είπε σήμερα ότι πρέπει ε, να υπάρχει σεβασμός ε, και γι' αυτό λέω σε εσά ντροπή σα. Ντροπή σα για αυτά τα επονίδη σχόλια που κάνατε. Ευχαριστώ κύριε Βιέγας. Θα ήθελα να εκφράσω την ελεγγύη μου και τη συμπαράστασή μου προς το λαό της Βενεζουέλας. Ο λαό με ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο εξέφρασε την υποστήριξή του στην επαναστατική διαδικασία που έχει ξεκινήσει στη Βενεζουέλα με την ε, μεγαλύτερη ε, ε, συμμετοχή σε εκλογές και την πιο αθρώα προσέλευση. Μάλιστα, ο Τζίμι Κάρτερ, πρώην ε, ε, πρόεδρος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ως υποδειγματική την εκλογική αναμέτρηση και τη δεξαγωγή των εκλογών στη Βενεζουέλα. Πριν δώσουμε μαθήματα δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ε, κρατικό πλούτο για να εξυπηρετήσει το κοινό καλό, να μειώσει την πείνα, τη φτώχεια, τον αναλφαβατισμό, ε, να δώσει στέγη σε όσους ζούσαν στο δρόμο. Ε, ε, πραγματικά έχει καταθέσει εναλλακτικά αναπτυξιακά σχέδια η Βενεζουέλα και νομίζω ότι η ιστορία θα κρίνει ποιος είναι δίκαιος και ποιος όχι. Ο κύριος Δελαβέντοβα. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ. Η Ευρώπη συνδέεται με ε, βαθιές, με βαθιές ιστορικούς δεσμούς με την Βενεζουέλα και πιστεύουμε ότι η Βενεζουέλα έχει την ε, δυνατότητα ε, να αποτελέσει κινητήρια ή τουλάχιστον θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη οικονομική και εμπορική για την, πολιτική, για την περιοχή. Επομένως μας προκαλεί μέγιστη ανησυχία αυτή η μεγάλη πόλωση ανάμεσα την στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Τον τελευταίο χρόνο είδαμε βίαιες διαμαρτυρίες. Ήδη από το Φεβρουάριο, μέσα από σειρά δηλώσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τη μεγάλη της ανησυχία για αυτήν την ισχυρή πόλωση και τον πολλαπλασιασμό των βιαίων επεισοδίων. Έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας όσον αφορά τον φυλακισμό ε, των πολιτικών ηγετών ε, καθώς επίσης και φοιτητών ε, που είχαν διαδηλώσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια συνενετική λύση. Καλέσαμε όλες ε, τις ε, πλευρές να φτάσουν σε πολιτική συμφωνία και οπωσδήποτε ε, να καταδικάσουν τη βία. Ε, δυστυχώς βλέπουμε ότι η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει. Αντιθέτως και για το μέλλον ε, προβλέπουμε τέτοιου είδους σενάρια αντιπαράθεσης. Εμείς είχαμε ήδη εκφράσει την συμφωνία μας με τα λεγόμενα του Προέδρου Μαδούρο τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του για τη δημιουργία ενός ενιαίου έθνου με άρση των εσωτερικών ε, διαφορών. Εμείς κάνουμε έκκληση στην αίσθηση ευθύνης ε, της κυβέρνησης αλλά και των άλλων εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να βρεθεί διέξοδος. Μονάχα μια ολοκληρωμένη λύση θα μπορέσει πραγματικά να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Θα πρέπει αυτά που είπε ο πρόεδρος Μαδούρο το 2013 να γίνουν πραγματικότητα. Να βρεθούν συνεργικές λύσεις για να προχωρήσει η χώρα προς το μέλλον. Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχουν μονάχα πολιτικά προβλήματα αλλά και προβλήματα οικονομικά ε, και ασφάλειας. Ε, ε, μία καταβαράθρωση της οικονομίας με αστρονομική, αστρονομικό πληθωρισμό, αύξηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας η μεγάλη μείωση παγκόσμια των τιμών του ε, πετρελαίου οπωσδήποτε βαραίνει στην ικανότητα της χώρας ε, να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της ανάγκες για το 2015. Αναγκάστηκε ο πρόεδρος ε, Μαδούρο να κάνει περικοπές όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση και το βάθεμα της κρίσης. Ε, ε, και η ευρύτερη περιοχή ενδεχομένως θα υποφέρει ε, από την κατάσταση αυτή όπως υπενθύμησε και πρόσφατα ο πρόεδρος της Μερκοσούρ ή πρόεδρος της Μερκοσούρ. Ε, η φυλάκιση των ε, ε, διαμαρτυρωμένων φοιτητών καθώς επίσης και των αρχηγών της αντιπολίτευσης θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ξεκινήσει αποτελεσματικές και αδέκαστες διερευνήσεις όλων των περιπτώσεων κατάχρησης. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτός ο δικαστικός αγώνας εναντίον ε, όλων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η πολιτική κράτηση όπως του Λεοπόλντο Λόπες και των φοιτητών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ενισχύσει τις σχέσεις της ε, με την Βενεζουέλα ε, και σε επίπεδο περιφέρειας και διμερός. Εμείς θέλουμε να δούμε σταθερότητα και πρόοδο στη Βενεζουέλα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ολοκληρωμένο διάλογο, σεβασμό Τη της ε, ελευθερίας έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ευρεία διαδικασία συμφιλίωσης. Ευχαριστώ. Με την ομιλία και το Συμβουλίου